ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και ήθελα να καλέσω τον κύριο Πυρίλο να μας παρουσιάσει την προφορική ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, από τη συνάδελφη να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνυπέγραψαν την προφορική αυτή ερώτηση. Στόχος ε, της ευρωπαϊκής προσπάθειας για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα και πολιτικές ε, που μπορεί να περιορίζουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ο στόχος περιορισμού των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα είναι ένας πολυμερής στόχος ώστε παρόλα αυτά ασκούνται πιέσεις στο ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύστημα, ιδίως στις ενεργοβόνες βιομηχανίες. Οι στόχοι που όλοι συμμεριζόμαστε στην, ε, στο σχεδιασμό τους θα πρέπει να, να επιδιώκεται να υλοποιούνται με τρόπο ρεαλιστικό. Θα πρέπει η Επιτροπή λοιπόν πιο συγκεκριμένα και με ακρίβεια να αναζητήσει τα κατάλληλα συστήματα εφαρμογής του συστήματος ανταλλαγής εκπομπών και τα μέσα χρηματοδότησης ώστε να εξορκίσει την έλλειψη ισορροπίας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός που τροποποιήθηκε το 2009 ε, προβλέπει από το 2013 οι ε, εταιρείε παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος να αγοράζουν ποσοστώσεις για το σύνολο των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή το μεγαλύτερο κόστος ε, θα μεταφερθεί στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και θα επιταθεί και το κόστος, θα αυξηθεί το κόστος ε, της παραγωγής. Γύρω στα τεκτιμά ότι το επιπλέον κόστος από το σύστημα αυτό που θα αυξήσει την τιμή του ρεύματος θα φτάσει 8,5 δις ευρώ ετησίως. Όμως δεν υπάρχει σύστημα αντιστάθμισης γιατί σε εταιρείε του ίδιου τομέα βλέπουμε διαφορετική μεταχείριση και πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών, δικαιωμάτων εκπομπών. Έτσι, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναζητήσουμε τη δημιουργία ενό συστήματο ισότιμου. Ιδάλω, θα έχουμε επαναγκατάσταση των εταιριών. Η επιλογή των τομέων που μπορεί να προκαλέσουν εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα είναι απλουστευτική. Θα πρέπει η παραγωγή ενεργοβόρων ε, ενεργειών να επιτραπεί εφόσον υπάρχουν και αντισταθμιστικά μέτρα. Για την παραγωγή ατσαλιού είναι δύο τα μέσα της παραγωγής. Η ηλεκτρική ε, φούρνη και τα ψυχρά και η ψυκάμινη οι υψικάμενοι θα υποφεληθούν από ποσοστώσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και αντιστάθμιση με την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό προκειμένου να μειωθεί η κομπή διοξιδίου του άνθρακα και βεβαίω και πάλι η παραγωγή αυτού του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σημαίνει και αυξημένο κόστος. Η αγορά αυτή επηρεάζει πολλούς βιομηχανικούς και βεβαίω εδώ πρέπει να δούμε και την απόκριση που σκέφτεται να δώσει σε όλα αυτά η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανία. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και να εξασφαλίσουμε ευημερία για του πολίτε. Πώ σκέφτεται όμω η Επιτροπή να συνεχίσει το σύστημα αυτό για τι ενεργοβόρε βιομηχανίε. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ισορροπίας που θα ε, δημιουργηθεί από το 2013 με τα σημερινά μέτρα δεν θα υπάρξουν τάσεις κερδοσκοπίας. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που θα προκληθεί. Ευχαριστώ. Πυρίλο, εξ ονόματος της Επιτροπής τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον Επίτροπο Σέμετα. Mrs. President, honorable members. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, Ξέρουμε μέλη, η Επιτροπή αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι το κόστος για την παραγωγή του χάλιβα και για την ε, επιρροή των κλιματικών αλλαγών στην διαμόρφωση τιμής του ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, συνειδητοποιούμε τις παρούσες οικονομικές δυσκολίες και την σημασία να υποστηρίξουμε με ευφυή μέτρα την οικονομική ανάκτηση και να δούμε πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε λιγότερο επικίνδυνες μορφές ενέργειας. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μία ευή ε, βιομηχανική, ε, βιομηχανία στην Ευρώπη, οι κρατικές ε, βοήθειες μπορούν να βοηθήσουν εάν κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές για να γίνουν με αηφόρο τρόπο αλλαγές στην βιομηχανία, αλλά δεν μπορούμε για κάποιους χρήστες μακροπρόθεσμα να εγγυηθούμε χαμηλότερο κόστος. Επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας σε μέτρα τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα, την δυνατότητα να κάνουν διαρθρωτικές βελτιώσεις στην βιομηχανία. Τα πλαίσια αυτής της οδηγίας, στα πλαίσια του πακέτου των κλιματικών λόγων του 2008, μπορούν να δώσουν αντισταθμιστικά ε, κονδύλια για το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στα κράτη ε, σε ε, βιομηχανίες και κυρίως να τους ενισχύσουν για τα θέματα της Η οικονομική αντισταθμίνοντα και η βοήθεια μπορεί όμως παρόλα αυτά γενικά στη γενική αγορά να δημιουργήσει στρεβλώσεις και να επιδεινώσει το σύστημα το οποίο ε, προβλέπεται για τα ε, θέματα της ε, ενίσχυσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται θα πρέπει η η οικονομική ενίσχυση να γίνεται στους τομείς ενεργομόνους γερίες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν χάσει ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουν, ε, έκαναν, μετεγκαταστάθηκαν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζοντας τις ε, κανόνες που πρέπει να ισχύουν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι απαραίτητες οι ενισχύσεις αυτές για να διασφαλίσουμε την ε, καλή υγεία της αγοράς. Αυτή τη στιγμή που έχουμε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και θα πρέπει να έχουμε ίσους όρους ανταγωνιστικούς για όλες τις βιομηχανίες του τομέα αυτού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα περάσουμε τώρα στους ε, ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ε, ομάδων και πρώτα θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Χέρμπετ Ρόιλ εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ ε, πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για τις δηλώσεις ε, της αρχής. Βεβαίως αυτές οι δηλώσεις δεν είναι απάντηση στην ερώτηση που σας έχει τεθεί, έτσι. Διότι οι ερωτήσεις τι θέλουν να καταλάβουν. Ε, είναι εξασφαλισμένο ότι θα έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα. Ε, θέλουμε οι βιομηχανίες να μην επιβαρύνονται τόσο πολύ ή να υπάρχει μια ε, ασφάλεια και αυτοί χρειάζονται ασφάλεια προγραμματισμού. Λοιπόν, γρήγορες αποφάσεις και σαφείς δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η διαδικασία τραβάει σε μάκρος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη και ο δρόμος που πήραμε, αλλά τότε, ε, αν θυμάστε, στην οδηγία για τα δικαιώματα εκπομπών ρήπων είχαμε πει ότι το κάνουμε ακριβώς υπό τον όρο ότι ενεργοβόρο χώρες βιομηχανίες στην Ευρώπη που θα επιβαρυνθούν ιδιαίτερα ε, θα μπορέσουν να ελαφρυνθούν αλλιώς θα χάσουν τον ανταγωνισμό με άλλους ε, γεωγραφικούς ε, τόπους. Και τότε ελήφθη αυτή η απόφαση στο Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και αναμένω να γίνει πραγματικότητα. Ανησυχώ λίγο ότι στο δρόμο χάνουμε τους δικαιούχους γίνονται όλο και πιο μικροί και κοντόφθαλμοι η προσέγγιση μας. Βγάζουμε απ' έξω όχι μόνο το χάλιβα, είναι και το αλουμίνιο, είναι η χημική βιομηχανία, δεν καταλάβαμε γιατί γίνεται αυτό. Και αυτό που ήταν πολιτική ε, βάση της απόφασης πρέπει να ελοποιηθεί. Σωστά είπατε κύριε Επίτροπε. Δεν διευκολύνθηκε η κατάσταση για την ευρωπαϊκή βιομηχανία από τότε που λήφθη η απόφαση. Δυσκολεύτηκε. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα ανταγωνισμού. Όλοι αγωνιζόμαστε και κηρύσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η βιομηχανία για το μέλλον της Ευρώπης. Εχθές ακούσαμε πάλι πολύ ευφυείς λόγους ε, το Κοινοβούλιο περιμένει, το, νομίζω ότι το περιμένει, αυτά που αποφασίσαμε να υλοποιηθούν σήμερα και μάλιστα προ όφελο εκείνων των κλάδων τη βιομηχανία που δεν είναι άνθρωποι και αυτοί που δουλεύουν, είναι θέσει απασχόληση, να έχουν και ευκαιρίε για το μέλλον στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόιλ. Εξ τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Μαρίτα Ούλσκοκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η βιομηχανία είναι καθοριστική για την ανάπτυξη τη Ευρώπη. Χωρί ανταγωνιστικότητα δεν θα προχωρήσει και ο τομέα των υπηρεσιών. Ε, αυτό είναι το θέμα ουσία, λοιπόν. Είναι σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι αυστηρότατη και να επαγρυπνεί και να είναι και ιδιαίτερα ενεργή όταν πρόκειται για θέματα ανταγωνιστικότητας ή πληγμάτων εναντίον της. Θα πρέπει λοιπόν να Έχουμε φιλοδοξίες λιγότερο υψηλές από την ε, περιβαλλοντική ενδεχομένως άποψη και θα πρέπει να υπερέχει και η δυνατότητα των εξαιρέσεων για κάποιους τομείς όπου υπάρχει εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά με τρόπο συνετό. Δεν δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να θεωρούμε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν θα αναλάβει τι ευθύνε τη. Σίγουρα θα επιδιώξει του στόχου τη ε, πολιτική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αλλά να θυμόμαστε ότι όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, απαιτείται δράση. Ε, έχοντας πάντα κατά νου τους στόχους των κλιματικών αλλαγών. Κατά καιρό μάλιστα Κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν τη σημασία τέτοιων παραγόντων και αυτό βέβαια έχει επιπτώσεις και στην αξιοπιστία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίζει αυτά τα αντιφατικά στοιχεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να έχουμε στόχους για να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω να ηγείται αυτή τη προσπάθεια. Χρειάζεται όμω ρεαλιστική προσέγγιση και να αναλύσουμε προσεκτικά τι αντίκτυπο έχουν τα μέτρα που παίρνουμε. Θα σταματήσουμε να δίνουμε δωρεάν άδειε. Αυτό θα έχει επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα ενεργοβόρων ε, κλάδων της βιομηχανίας. Βεβαίως η βιομηχανία πλήττεται με διαφορετικό τρόπο, όπως είπε και ο κύριος Πυρίλο, ανάλογα με το είδος της. Στη Ρουμανία, Φέρυπιν, ο μισός χάλιβας παράγεται σε ηλεκτρικές υψηκαμίνου και θα έχουμε μεγάλο αντίκτυπο. Αντίστοιχα ισχύουν και σε άλλα κράτη-μέλη. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η αγορά του χάλιβα είναι παγκόσμια και ε, ο περιορισμός των εκπομπών είναι καλός στόχος αλλά κινδυνεύει να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό. Αν δεν υπάρχει παγκόσμια συμφωνία προς την κατεύθυνση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δει τη βιομηχανία της να πιέζεται, να πλήττεται. Γι' αυτό κινδυνεύουμε να σηκωθούν και να φύγουν οι βιομηχανίες. η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές της μελλοντικέ για τις ε, κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να πει ότι 24 ε, Δεκεμβρίου 2008 ελήφθη μια απόφαση που θα πρέπει να ισχύει για όλους, για το έμεσο κόστος του ETS, του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρήπων. Αλλιώς είναι η μη μέτρα αυτά που παίρνουμε και ε, διακυβεύουν την ανταγωνιστικότητα και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μειώνονται και εκπομπές παγκοσμίως. Ευχαριστώ. των Ευρωπαίων Συντηρητικών, ο κύριος Σιμάνσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Panie komisarzu, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, λόγω της πολιτικής καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών, οι ενεργοβόρες βιομηχανίες μας δέχονται τεράστιες πιέσεις, ε, ιδίως στην ανταγωνιστικότητά τους και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχουν όρια εκπομπών, σκεφτείτε την βιομηχανία, τη χημική, της παραγωγής χάρτου, του χαλιβουργία. Θα υπάρξουν λιγότερες επενδύσεις, λιγότερη καινοτομία και μετεγκαταστάσεις ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι βιομηχανίες αυτές ε, έχουν και δυσανάλογο κόστος στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ακριβώς ε, γιατί χρειάζεται να εκπέπεται άνθρακας για να υπάρχει παραγωγή όπως και το χάλιβα και αυτό συμβαίνει και στην Πολωνία. Αν δεν θέλουμε λοιπόν να χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας πρέπει να διευκολύνουμε τους τομείς αυτούς ώστε να μπορέσουν να περάσουν σε μεθόδους παραγωγής με μικρότερη εκπομπή άνθρακα αλλά με μέτρα στηρίξης και προστασίας. Ε, της ομάδας Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κύριος Ρώση, για ένα λεπτό παρακαλώ. Συνάδελφοι, και στην Επιτροπή μας και εδώ στην Σύνοδο Λομέλειας κατήγγυλα ότι μπορεί τα μέτρα αυτά να γίνουν ε, αφορμές για κερδοσκοπία και πολλέ χώρε να μετακατασταθούν σε τρίτες χώρες γιατί δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ο αντίκτυπο ε, των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα που θα μεταφερθεί στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πλήξει το μηχανικό σύστημα κατά τρόπου διαφορετικούς. Οι τομεί που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια όπως τη χαλιβουργίας και της παραγωγή αλουμινίου, της ερασματοπίας θα γνωρίσουν αυξημένο κόστο. Θα πρέπει λοιπόν ε, το κόστο αυτό να, μην το επομίζονται μόνο του εταιρείε των κρατών μελών. Θα πρέπει για να αναχαιτήσουμε τον κίνδυνο των μετακαταστάσεων να λάβουμε μέτρα. Επίση, η οικονομική αποζημίωση, ακόμη και για την ενέργεια που καταναλώνεται, ε, δεν θα πρέπει να είναι κάτι που να μας απασχολήσει. Και για λόγους γραφειοκρατικούς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες ε, ε, θα έπρεπε να υπάρχουν ενισχύσεις ή μήπω θα υπάρξει έτσι στρέβλος του ανταγωνισμού σε σχέση με εταιρείε σε τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, τελευταία εγγεγραμμένη ομιλήτρια, η κυρία Ντότζ από τους μη εγγεγραμμένους, αλλά δεν την βλέπω στην αίθουσα. Οπότε θα περάσουμε στους ε, υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Λίζε. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίλο που έφερε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Διότι δεν έχουμε εμεί άμεσε μεν αρμοδιότητε για το θέμα, αλλά θα πρέπει να πιέσουμε λίγο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα δεν είναι μόνο η ηλεκτρική παραγωγή χάλιβα. Το είπε και ο κύριος Ρόιλ. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι, το αλουμίνιο και η χημική βιομηχανία που κινδυνεύουν να μετασταθούν οι επιχειρήσει θα πρέπει να ενταχθούν, οφείλουν να ενταχθούν σε αυτές τις ενισχύσεις και τονίζω το οφείλουν γιατί το λέει και η οδηγία. Το θέμα μας, το πρόβλημά μας δεν είναι η οδηγία. Ούτε χρειάζεται να αλλάξει. Ε, ισχύουσα μέχρι το 2011 δεν περιλαμβάνει αυτή τη ρυθμίση, αλλά στη νέα ορίζεται ρητά ότι ε, ε, και στις άμεσες και στις έμεσες εκπομπές χρειάζεται υποστήριξη. Γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει να ελοποιήσει αυτά που έχουμε αποφασίσει. Το πρόβλημα δεν είναι το κείμενο τη οδηγία, που θα έλεγα ότι είναι και καλύτερο γιατί έχουμε τη δυνατότητα αποζημίωση που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ανασκουμποθεί και χρειαζόμαστε ένα σαφές πλαίσιο ενισχύσεων με διαφάνεια. Αλλιώς έχουμε κρυφές επιδοτήσεις σε διάφορα κράτη-μέλη και τότε είναι που στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. Το λέω ξεκάθαρα. Ορισμένες επιχειρήσεις περιμένουν, δημονούν, χάνουν ήδη από σήμερα ή τουλάχιστον δεν κερδίζουν διότι τα πιστοποιητικά και οι άδειες ακόμα και αν μοιράστηκαν δωρεάν ε, τώρα έχουν ε, συμπεριληφθεί στην τιμολόγηση. Αν δεν δουν λοιπόν φως στο τέλος του τούνελ ε, από το 2013 ότι θα έχουν ενισχύσει αυτές οι εταιρείε, ενδεχομένως να λάβουν αποφάσεις που δεν θα μας αρέσουν στην Ευρώπη ως τόπο παραγωγής. Βεβαίω δεν θα πρέπει να υπάρξει υπερβολική αποζημίωση, αλλά ούτε υποαποζημίωση και θα πρέπει πάντα να τονίζουμε ότι έχουμε και benchmarks, έχουμε συγκριτική αξιολόγηση. Πρόκειται για τι 10% καλύτερε εταιρείε και αυτό είναι αρκετό κίνητρο να είσαι αποτελεσματικό και παραγωγικό, και τώρα καλύτερα να το εφαρμόσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σεντσιου για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η χαλιβουργία αποτελεί τη βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πυλώνες της βιομηχανίας της. Ε, χωρίς τη χαλιβουργία δεν μπορούμε στην Ευρώπη να διατηρήσουμε την ανάπτυξη, την παρουσία μας στην παγκόσμια αγορά. Η παγκόσμια αγορά, ξέρετε, δεν έχει δεσμευτικούς κανόνες. Η χαλιβουργία και η βιομηχανία ε, αλουμινίου καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν έχουμε στόχους για τη μείωση των εκπομπών, ε, θα αυξηθεί μοιραία η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η χαλιβουργία και ε, η βιομηχανία του αλουμινίου χρειάζεται όμως ηλεκτρικές υψηκαμίνους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό ε, και να τους δοθούν δωρεάν άδειες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική παγκοσμίω και να ε, μην έχει μειονεκτήματα απέναντι σε ε, εργοστάσια κρατών που επιδοτούνται. Κυρία Κόμη, για λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το θέμα μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ, επειδή μια τέτοια οδηγία μπορεί να έχει σοβαρό αντίκτυπο για του ε, τομεί που είναι ενεργοβόροι στη βιομηχανία. Οι προθέσει μα αυτέ να κάνουμε το σύστημα πιο αποτελεσματικό μπορεί τελικά να επηρεάσουν την έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε να επωφεληθούν οι εταιρείε και όλο ο τομέα και από την αύξηση τη παραγωγικότητα και βεβαίω από την ε, καινοτομία. Επίση, να μην ξεχνάμε ότι σημαντικό είναι το τι θα συμβεί και με την απασχόληση. Δεν θέλουμε να υπάρξει διακριτική μεταχείριση μεταξύ διαδικασιών και εταιρεών ώστε να μεταγκατασταθούν εταιρείε εκτό Ευρώπη και να χαθούν εταιρείε που δίνουν θέσει εργασία, που αποφασιστικά συμβάλλουν στην παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση του πλούτου στην Ήπειρο. Ε, η αγορά εργασία και παραγωγικότητα, καθώ και επένδυση στι ε, ανακυκλώσιμε πηγέ ενέργεια, είναι καθοριστικοί πυλώνε για την οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ανάπτυξη τη Ευρώπη. Ήθελα να σταθώ στην ανάγκη να αποφύγουμε ε, την αύξηση του κόστου για τι εταιρείε που μπορεί να δημιουργηθεί στρέβλωση στην ανταγωνιστικότητα τη αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ροβάνα Πλούμπ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει κάποια αλλαγή για αυτές τις ενεργοβόρες βιομηχανίες χρησιμοποιώντας ε, πιο ανταγωνιστικές ε, ε, μεθόδους θα πρέπει να μειωθεί η εκπομπή ρίων και να χρησιμοποιούν ευφύς μηχανισμοί για να διατηρηθούν οι παρούσες ε, καλύτερες πρακτικές. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ε, κάτι για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικές οι εταιρείες αυτές, διαφορετικά θα χάσουν την ε, ανταγωνιστικότητά τους με το θέμα της μεταφοράς των δικαιωμάτων εκπομπής και θα χαθούν νέες επασχόλησεις. Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βον Ρόι, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η πολιτική για το διοξίδιο του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυναμική ε, ε, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για τους ευαίσθητους τομείς. Τώρα έχουμε ένα κόστος ε, της ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο μετακυλίεται σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, χαλιβουργία, αλουμίνιο και χημική βιομηχανία. Αλλά δεν θα πρέπει να ε, είναι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας αυτών των εταιριών. Το θέμα είναι στη μετακύληση του εμέσου κόστους από την ηλεκτρική ενέργεια ε, στις βιομηχανίες. Αυτό που μας χρειάζεται κύριε Επίτροπε είναι καλή πληροφόρηση, ευρύτατη σε όλη την Ευρώπη για το άρθρο 10 το οποίο δεν είναι τυχαίο ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να μην έχουμε πάλι άνισους κανόνες παιχνιδιού. Θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια για όλες τις εταιρείες στην Ευρώπη και μάλιστα ε, γρήγορα. Και μια ερώτηση. Η Γερμανία εγκαταλείπει την ατομική ενέργεια. Αυτό τι επιπτώσεις έχει, ε, μεγάλες επιπτώσεις ε, σε αυτό τον κλάδο. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλσίτης για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Πυρίλο, που θέσατε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Οι δεσμευτικέ, ε, οι δεσμεύσει μάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών μα υποχρεώνουν να κάνουμε την βιομηχανία μα πιο πράσινη, να περάσουμε σε έναν δρόμο πιο οικολογικό. Όμω εδώ μπορεί να υπάρχει και αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένου βιομηχανικού τομεί που καταναλώνουν ιδιαίτερε υψηλέ ποσότητε ηλεκτρικού ρεύματο. Και πολλέ εταιρείε μπορεί να χάσουν την ε, ανταγωνιστικότητά του εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κίνα, λόγω χάρη έχει το ευρύτερο δίκτυο χαλιβουργία παγκοσμίω και τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει προσεκτικά και υπεύθυνα να εξετάσει τα ζητήματα αυτά σε σχέση με τι κρατικέ ενισχύσει και να βρει μια σωστή ε, ισορροπία μεταξύ των δεσμεύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα πλεονεκτήματα τη ανταγωνιστικότητα τη αγορά μα από τα οποία εξαρτάται η ανάπτυξη και η ευημερία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τώρα τη προφορική ερώτηση, ο έχει λεπτό. Παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις που πήραν το λόγο και ενίσχυσαν την ερώτησή μου. Δεν μπορώ να πω ότι ικανοποιήθηκα πλήρως, διότι είχαμε και το ΚΑΤΣΤΙΑΙ. Και θα πρέπει να ακούσουμε τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ σαν να υπάρχει μια αντίφαση. Ελπίζω ότι οι διαδικαστικοί κανόνε θα προσαρμοστούν για να λυθεί και αυτό. Πάντω, μέσω του τύπου θα μπορέσω να συμπλώσω την απάντησή μου, όμως απογοητεύομαι, απογοητεύομαι από την απόκρισή σα Επίτροπε, στη συγκεκριμένη αυτή ερώτηση. Δεν νομίζω ότι θέλει να φαίνεται ότι είναι υπτητας χείρας στη η Επιτροπή. Έτσι βέβαια το εξέλαβαν οι συνάδελφοι και ελπίζω ότι η Επιτροπή στο γραπτός θα απαντήσει στην ερώτησή μου. Ελπίζω ότι θα εξετάσετε σοβαρά το σοβαρότατο αυτό το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω δύο συναδέλφους ε, ε, στην ε, λίστα και πρώτα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιασλοβιέσκα. Δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Σίλβια Τσικάο να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Εγώ είμαι από το Γαλάτσι. Ξέρετε, είναι μια πόλη που έχει μεγάλη και χαλιβουργία και ε, ναυπηγική βιομηχανία. Και η χώρα μου και η περιοχή μου εξαρτάται κατά πολύ από τις βιομηχανίες αυτές και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, που επιτρέπει να ε, δρούν αυτέ οι βιομηχανίε. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οι θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε τις ενεργοβόρε βιομηχανίες. Κάνουμε συζητήσεις για τι άδειε εκπομπών ρήπων ε, για τι βιομηχανίε αυτέ, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ευνοϊκούς όρους για τις εταιρείες αυτές που επενδύουν σε πιο πράσινη τεχνολογία και σε πιο ε, μεγάλη εξοικονόμηση και αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Η ίδια η επιβίωση της βιομηχανίας μας θα εξαρτηθεί από τα μέτρα που τώρα λαμβάνουμε για να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι εταιρείε και μιλώ ιδιαίτερα για τη Χαλβουργία. Ευχαριστώ. Τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής να παρακαλέσω τον Επίτροπο Σέμετα Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Πυρίγιο για την ερώτηση που υπέβαλε και θα ήθελα να πω με σαφήνεια ότι η Επιτροπή δεν είναι τα σχήρες της για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Είπα με σαφήνεια ότι οι σε επιπτώσου για τις κρατικέ συνεχίσεις που δίδουν σε αυτές τις ενεργοβόρες βιομηχανίες συνεχίζεται και αυτή η ε, ανάλυση επιπτώσεων περιλαμβάνει τη χαλιβουργία και άλλες βιομηχανίες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Άρα, σήμερα αν δεν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη επιπτώσεων, δεν μπορούμε να καταλύσουμε σε οριστικά συμπεράσματα για το ποιοι τομείς της βιομηχανίας θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των καθευθυντήριων γραμμών. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, η πρόθεση της Επιτροπής είναι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές μέχρι το τέλος του έτους να ε, εγκριθούν μετά από δημόσια διαβούλευση. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έστειλε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο για τα αμφιλεγόμενα σημεία για την ε, ε, δικαιούσους σε ε, κοινοτικό επίπεδο. Έχουμε πάρει 140 ερωτήσεις από τη βιομηχανία, από διάφορες υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και αναλύουμε τις απαντήσεις και μετά θα κάνουμε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χορήγηση αυτών των κρατικών ενισχύσεων. Τα κράτη-μέλη θα τα συμβοληφτούμε κάποια άλλη χρονική στιγμή πριν να κάνει έγκριση κάποιων αποφάσεων η Επιτροπή και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί. Η όλη διαδικασία είναι διαφανής και θα προβούμε στις προτάσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες ως το τέλος του έτου. Η συζήτηση γύρω από την προφορική αυτή ερώτηση ολοκληρώθηκε και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι δήλωση της ε, Επιτροπής για τους ε, Σαρωτές Ασφαλείας. Θα ήθελα και πάλι να παρακαλέσω τον ε, Επίτροπο Σέμετα, εξ ονόματος της Επιτροπής.